τίτλοι θα δημοσιευτούν στα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης. Περνάμε τώρα στην έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Όπως αυτή είχε εγκριθεί και την έχετε λάβει. Για την Δευτέρα το ΕΛΚ μου ζητάει πώς θέλει η συζήτηση για την ε, για την πρόταση της Κομισιόν για τις οδηγίες αξιολόγηση αντικτύπου θέλει να καταλήξει σε ένα ψήφισμα. Δίνω τον λόγο στον κύριο Πίπερ για να αιτιολογήσει το αίτημα αυτό του ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απόψε θα συζητήσουμε το θέμα των ε, μελετών επιπτώσεων, δυστυχώς ε, χωρίς ε, κάποιο ψήφισμα και μιλάμε για τις επιπτώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, που δυστυχώς πλέον δεν ε, θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στην νέα πρόταση της Κομισιόν. Οι γενικοί διευθυντές ε, δυστυχώς εκμεταλλεύονται το περιθώριο εκείνο το οποίο έχουν και άρα δεν θα λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν θέλουμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο, γι' αυτό ζητάμε ένα ψήφισμα μετά από την συζήτηση αυτής της εβδομάδας και ζητάω την στήριξή σας. Σας ευχαριστώ. Θέλει κάποιος να στηρίξει τον κύριο Πίπερ, παρακαλώ. Πρόεδρε, σύμφωνο με την πρόταση το κείμενο βεβαίω του ψηφίσματο πρέπει να συζητηθεί. Είμαστε μακριά ακόμη από το να καταλήξουμε στο τελικό κείμενο, αλλά το υποστηρίζουμε. Σα ευχαριστώ. Θέλει κάποιο να τοποθετηθεί κατά. Κατά. Κανεί. Ωραία. Θα το ψηφίσουμε. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λοιπόν, οι προθεσμίες είναι εξής. Για προτάσεις ψηφίσματος 3η 12 η ώρα, για τροπολογίες και κοινά ψηφίσματα 12 η ώρα Τετάρτη, τροπολογίες επί των κοινών ψηφισμάτων 1 η ώρα Τετάρτη. Για χωριστές ψηφοφορίες Τετάρτη 7 το απόγευμα. Η δε ψηφοφορία θα λάβει χώρα την 5η για την Δευτέρα. Υπάρχουν άλλα αιτήματα αλλαγής και διάταξης. Όχι. Για την Τρίτη. Το ΕΛΚ έχει ενημερώσει πως θα ήθελε να αποσυρθεί το αίτημα για ψήφισμα για την γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την ανταλλαγή δεδομένων με ΗΠΑ και Καναδά, τα λεγόμενα PNR. Η κυρία Χόλμαϊρ έχει πρώτα απ' όλα το λόγο για να αιτιολογήσει το αίτημα αυτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το αίτημα αυτό υπευλήθη πριν από τρει ημέρε ε, χωρίς να συνοηθούν οι συζητητές. Γι' αυτό οι ομάδε δεν, δεν είχαν την ευκαιρία να το συζητήσουν ούτε καν στην Επιτροπή δεν έχει γίνει κάποια συζήτηση εις βάθος. Θεωρώ πως είναι αναγκαίο να έχουν χρόνο οι Επιτροπές να το συζητήσουν. Είναι προβληματικό επίσης όταν μιλάμε για διεθνείς ε, συμφωνίες να δίνουμε τέτοια άσχημη εικόνα γιατί αποδεικνυόμαστε μη αξιόπιστοι εταίροι. Και βεβαίως το να λαμβάνονται πολιτικές ε, αποφάσεις ε, προδικάζοντας ε, την οριστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι λάθος. Τίθενται ζητήματα νομικής ασφάλειας για τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες. Οπότε βρισκόμαστε σε ένα δύσκολο και ευαίσθητο θέμα όπως η καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας η οποία κινδυνεύει να πάει πίσω από 12 μέχρι 36 μήνες γιατί δεν μπορούμε να δράσουμε παρκώς. Σας ευχαριστώ. Ποιος θέλει να υποστηρίξει την κυρία Ολμάιρ υπέρ. Ποιος. Ναι, ναι, το αιτιολογήσατε, ε, μπορεί και... Μάλιστα. Κατά, κάποιος θέλει να επιχειρηματολογήσει, κυρία Ζίπελ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γιατί είμαστε εμείς υπέρ της ε, προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ποτέ δεν είχε αμφισβητήσει πώς οι αεροπορικοί επιβάτες μπορεί να είναι ένα στοιχείο καταπολέμησης τρομοκρατίας και είχαμε συμφωνήσει σε δύο συμφωνίες στο παρελθόν, αλλά αυτό το κάναμε σε μια φάση κατά την οποία η αποθήκευση των δεδομένων ήταν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τω μεταξύ όμως αυτή η οδηγία από ό,τι φαίνεται κατέπεσε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Πρόκειται για την πρώτη διεθνή συμφωνία που θα αποφασίσουμε μετά από αυτή την απόφαση και οπωσδήποτε οι διαπραγματευτέ δεν θα το ξεκαθαρίσουν αυτό στι διαπραγματεύσει. Αλλά θα ήθελα να επενδυμίσω πω Συμβούλιο και Κομισιόν πρέπει να ξεκαθαρίσουν το κατά πόσον αυτή η μορφή των δεδομένων αεροπορικών επιβατών είναι συμβατή με τις ευρωπαϊκές συνθήκες, κάτι το οποίο δεν έκαναν. Κίνδυνος για τους πολίτες ε, Ευρώπης και Καναδά δεν βλέπω εγώ να υπάρχει. Κρατάνε πέντε χρόνια οι διαπραγματεύσεις ρέουν τα δεδομένα και θα συνεχίσουν να ρέουν. Νομίζω πως είναι μια καλή παράδοση το να σιγουρευόμαστε ότι αυτά τα οποία κάνουμε για την ασφάλεια των πολιτών μας δεν παραβιάζουν τα θεμελιώδη τους δικαιώματα. Θα ψηφίσουμε. Ποιος είναι υπέρ του αιτήματος της κυρίας Χολμαέρ να φύγει το θέμα από την ημερήσια διάταξη κατά αποχές απορρίπτεται. Καλώς. Να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Ε, εντάξει, τι να σας κάνω. Ψήφισαν όλοι. Ε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα μα αργείτε τόσο. Απορρίπτεται το αίτημα. για την Τρίτη. Θέλει κάποιο κάτι άλλο επί τη ημερήσια διάταξη. Όχι, Τετάρτη. Το ΕΛΚ ζήτησε αναβολή της ψηφοφορίας ε, του ψηφίσματος για την αναγνώριση του κράτους της ε, Παλαιστίνης για το Δεκέμβριο. Ο κύριος Πρέντα έχει το λόγο. Πρόεδρε, εκ μέρους του ΕΛΚ ζητούμε την αναβολή της ψηφορίας για αυτό το λεπτό θέμα. Πιστεύω ότι η συζήτηση μπορεί να γίνει όπως προγραμματίσαμε και καθώς ε, θα έχουμε περισσότερο χρόνο μπροστά μας, ψηφίζουμε τον Δεκέμβριο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε προς τα έξω την εντύπωση ότι είμαστε διηρημένοι σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Είναι κάποιο υπέρ του του κύριου Πρέντα. Κατά. Παρακαλώ κύριε Χάουιτ. Πρόεδρε, σύμφωνα με τα όσα είπατε για τη συναγωγή και την επίθεση, την τρομερή αυτή επίθεση. Δεύτερον, για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε να ψηφίσουμε αλλά να είμαστε ενωμένοι. Τουλάχιστον να εξασφαλίσουμε μια μεγάλη πλειοψηφία. Το ζήτησαμε και με τον κύριο Πρέντα. Το ΕΛΚ δηλώνει ότι είναι σταθερό στη θέση του, δεν θα κάνει υποχωρήσει. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε όμως βήματα, αλλά Γι' αυτό χρειάζονται συνομιλίε, διαπραγματεύσει. Αν δεν προσπαθήσουμε όλοι, δεν πρόκειται να φτάσουμε πουθενά. Να πούμε ότι το Παλαιστινιακό κράτο είναι μια συμβολή σε μια λύση με δύο κράτη. Να πούμε ότι υποστηρίζουμε τη διαδικασία διαπραγμάτευση κλπ. Μπορούμε να βρούμε λοιπόν μια συμβαστική λύση, αφού μιλήσουμε όμω. Δυστυχώ όμω το ΕΛΚ δεν βλέπω να αποζητά τέτοια συμβαστική λύση. Γι' αυτό θα ήθελα να καλέσω όλους να μιλήσουμε για το κείμενο σε αναζήτηση συμβαστικής λύσης. Και επίση θέλουμε να είμαστε συμμέτοχοι στην διαδικασία στη Μέση Ανατολή ή όχι. Θα ψηφίσουμε τώρα το αίτημα το αίτημα αναβολής για τον Δεκέμβριο. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι οι συνάδελφοι. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. 188 υπέρ. 167 καταγίνεται δεκτό το αίτημα. Επίσης για την Τετάρτη η Ευρώπη της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας ζήτησε να αλλάξει ο τίτλος ε, της δήλωσης Κομισιόν για τον Χάλιβα. Ο κύριος Ταμπουράνο έχει το λόγο. Χαίρετε. Λόγω τη σημασία του θέματο όσον αφορά τι κοινωνικέ και επαγγελματικέ πτυχέ και το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση γεννήθηκε αρχικώ ω κοινή αγορά άνθρακα και χάβυλα ε, χάλιβα εξ του EFTD, ε θα θέλαμε ε, την Τετάρτη να έχουμε τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την Ευρωπαϊκή ε, Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα να αλλάξει και να είναι τομέας της χαλιβουργίας προστασία των εργαζομένων και να έχουμε τη δυνατότητα ψηφίσματος το οποίο θα ψηφιστεί το Δεκέμβριο για να έχουμε απαραίτητο χρόνο για να διαπραγματευτούμε το ψήφισμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Είναι κάποιος υπέρ. Κατά. Ωραία, να το ψηφίσουμε. Ποιο είναι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Το αίτημα γίνεται δεκτό. Επίσης την Τετάρτη, οι Ευρωπαίοι συντηρητικοί και μεταρρυθμιστές συζήτησαν δήλωση από την Κομισιόν για τις παρατυπίες στις δημοτικές εκλογές της Πολωνίας και τον κίνδυνο για την δημοκρατία να προσθεθεί ως τελευταίο θέμα Τετάρτη βράδυ με ψήφισμα. Ποιος θέλει να στηρίξει αυτό το αίτημα. Ο κύριος Κρασνοντεύσκη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε, θα ήθελα και ζητώ να συμπεριλάβουμε στη μέση διάταξη αυτό το οποίο μόλις είπατε. Πρόκειται για εξόφθαλμες παρατυπίες, ανομαλίες που διαπιστώθηκαν στην Πολωνία πρόκειται για μια απειλή κατά της δημοκρατίας. Η πιο σοβαρή από το 1989. Ζητώ λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, δήλωση της Κομισιόν επί του θέματος ε, μαζί με συζήτηση. Οι εκλογές που λέμε χώρα στην Πολωνία δεν συνάδουν με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα. Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι συνέβησαν σοβαρές παρατυπίες. Στην Πολωνία ξεσκόθηκε γενική καταγραφή. Τα αποτελέσματα, να φαρεστείτε δημοσιεύτηκαν έξι ολόκληρε μέρες μετά από τις εκλογές. Και εν μεταξύ είχαν ξεσπάσει διαμαρτυρίε ανά την Πολωνία από ανθρώπους που είναι πεπισμένοι ότι όντω συνέβησαν τέτοιου είδου παρατυπίε. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολούμεθα πολύ συχνά με θέματα δημοκρατίας, και διαδικασιών και δημοκρατικών διαδικασιών. Να κοιτάζουμε όμως τι γίνεται και στον οίκο μας, όχι μόνο έξω. Ευχαριστώ κύριος Λεγκούτκο. <coughs> Uh, Κυρίες και κύριοι, έχω εδώ τα πρότυπα του ΩΣΑ, τα κριτήρια αν θέλετε, περί δημοκρατικότητας των εκλογών. Αυτά τα οποία συνέβησαν στην Πολωνία όντως παρεμβαίνουν τα πρότυπα αυτά. Όμως, κύριοι, αυτά συμβαίνουν στη χώρα σας. Πολλές φορές μετρήθηκαν 20% ή και 40% άκυρα ψηφοδέλτια. Για φαραστήρια αυτά να γίνονταν στη χώρα σας, να παρετούνται ολόκληρες εκλογικές επιτροπές. Αυτό εσείς, κατά τη γνώμη σας, θα το βρίσκετε συμβατό με τους δημοκρατικούς θεσμούς και τις δημοκρατικές διαδικασίες. Αν ναι, τότε να καταψηφίσετε. Εάν θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα, παρακαλώ να μας υποστηρίξετε. Θέλει κάποιος να τοποθετηθεί κατά του αιτήματος κ. Σόλμπρικ. Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, είμαι κατά του ψηφίσματος. Πρόκειται για απόπειρα εισαγωγής ε, τοπικών πολιτικών ζητημάτων στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για μια εσωτερική πολιτική υπόθεση. Τόσα συνέβησαν, πιστεύω και εγώ, όντως ε, ήταν μια αστοχία συστηματών πληροφορικής, ε, αστοχία ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συστημάτων κλπ. Αυτή τη στιγμή ανεξάρτητα δικαστήρια εξετάζουν τις λεπτομέρειες. Για όλους αυτούς τους λόγους προτείνω να καταψηφίσουμε το ψήφισμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε ποιο είναι υπέρ του αιτήματος αυτό κατά αποχές απορρίπτεται ε, σαφώς, για την πέμπτη δεν έχω κάποιο αίτημα οπότε οριστικοποιήθηκε η ημερήσια διάταξη τώρα περνάμε στο σημείο που λέγεται πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής. Να υπενθυμίσω το εξής. Σε αυτή τη συζήτηση δεν υπάρχει και HDI ούτε μπλε κάρτες. Καλωσορίζω πρώτα απ' όλα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που από ό,τι βλέπω είναι εδώ πέρα σύσσωμη πλην του κυρίου